σοβαρά υπόψη. Να είστε καλά. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε. Σας ευχόμαστε για τις ευθύνες ε, που αναλαμβάνετε. Καλή επιτυχία και ελπίζουμε να έχουμε και καλή συνεργασία. Τελειώνει λοιπόν εδώ η συζήτηση για το πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης την προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Κομισιόν. Να υπενθυμίσω σε όλους τους βουλευτές πως σε αυτό το θέμα δεν υπάρχει διαδικασία KCI. Μόνο ομιλητές των κοινοβουλευτικών ομάδων και ξεκινάει η συζήτηση από τον ε, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Σεύκοβιτς. Really... Ε, πρόεδρε, κύριε και κύριοι βουλευτές, ε, χαίρομαι ιδιαίτερα για τη σημερινή συζήτηση γιατί έρχεται σε μια κέρια στιγμή. Πρέπει να θυμόμαστε πως μόνο δύο χρόνια απομένουν για την θητεία αυτή του Κοινοβουλίου και θα συνεχίσουν να είναι στιγμές κρίσιμες για τους Ευρωπαίους, για τις δουλειές τους και για τις ευρωπαϊκής κοινότητας και θα πρέπει βεβαίως ε, να διασφαλίσουμε την αντοχή του οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου μας. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση απέδειξε πως είναι ένας απολύτως απαραίτητος παίκτη στην αντιμετώπιση της κρίσης. Αυτό μαζί όλοι δώσαμε στοχευμένες λύσεις στις ε, κατεπίγουσες κρίσεις και είδαμε βεβαίως και τις μακροπρόθεσμες προκλήσεις. Επίσης δώσαμε βάρος σε μια νέα οικονομική διακυβέρνηση, αναδιαμορφώσαμε όλο το σύστημα εποπτείας ε, του χρηματοπιστωτικού τομέα και βεβαίως η στενή συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων έχει ήδη αποδώσει. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε με τη σωστή ισορροπία μεταξύ υγιών δημοσίων, δημοσίων οικονομικών και επιτυχημένων επενδύσεων. Έτσι λοιπόν σκοπεύουμε να προωθήσουμε μια φιλόδοξη συμφωνία για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο κατά το κρίσιμο για να έχουμε ανάπτυξη και δουλειές. Έτσι θα έχουμε μια στέρεη βάση καθώς προσπαθούμε να ορίσουμε τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης τα επόμενα χρόνια και πάνω σε αυτήν μπορούμε να οικοδομήσουμε συγκεκριμένες Συγκεκριμένα ψηφίσματα των ομάδων υπογραμμίζουν το ότι υπάρχει ευρεία συνένεση σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα και σε όλα τα θεσμικά όργανα για το πώς η ευρωπαϊκή διάσταση μπορεί να κάνει τη διαφορά σε καιρούς μεγάλης οικονομικής δυσκολίας. Επίσης, είναι σημαντική ένδειξη του ότι συγκλίνουν οι προτεραιότητες μας, το ότι πολλές προτεραιότητες ε, του Κοινοβουλίου έχουν αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασία της Κομισιόν και προβλέπεται να υιοθετηθούν από την Κομισιόν αργότερα φέτος. Στην συζήτηση για την κατάσταση της Ένωσης που θα γίνει στις 12 Σεπτεμβρίου και έγινε πέρσι με στις 12 Σεπτεμβρίου παρουσίασε τις ε, βασικές προτεραιότητες μας ο πρόεδρος Μπαρόζο και το ίδιο θα κάνει και φέτος. Αυτές θα είναι η οικονομική ανάκαμψη και οι δουλειές με βάση στρατηγική του 2020 και είδαμε στο ευρωπαϊκό εξάμεινο πως η στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 και οι στόχοι της ενσωματώνονται στις ε, συστάσεις αναχώρα και στα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα όπως πολύ καλά γνωρίζετε ολοκληρώθηκε μόλις το δεύτερο ευρωπαϊκό εξάμεινο και οι άνα χώρα δίνουν ξεκάθαρες κατευθύνσεις στα κράτη-μέλη για εθνικές μεταρρυθμίσεις για δουλειές και ανάπτυξη μέσω και μακροπρόθεσμα. Και το ευρωπαϊκό επίπεδο τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να έχει ως στόχο να συμπληρώσει αυτές τις προσπάθειες εκεί πέρα ακριβώς όπου υπάρχει υψηλή προσθέμενη κοινοτική αξία. Μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της προηγούμενης εβδομάδας μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να κινηθεί αποφασιστικά σε μια νέα φιλόδοξη φάση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και αυτή είναι σαφώς η σωστή επιλογή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάτι το ενθαρρυντικό εν ώψη των πρωτοφανών προκλήσεων. Βεβαίως, για να είναι επιτυχές κάτι τέτοιο πρέπει πρώτα απ' όλα να βασίζεται στην κοινοτική μέθοδο και να έχει την πλήρη στήριξη του Κοινοβουλίου. Same time. Ταυτόχρονα πρέπει να διατηρηθεί η διαδικασία ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς για να υπάρξει το καθένα περιβάλλον για βιομηχανίες και υπηρεσίες, να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική χρήση των πόρων και την αηφορία, να έχουμε καλύτερη βιομηχανική πολιτική, να έχει ο κόσμος καλύτερη εκπαίδευση και δεξιότητες, να προωθήσουμε τα δικαιώματα των πολιτών και βεβαίως ένα θετικό αντίκτυπο στον κόσμο. Πάντα η Ευρώπη οικοδομείται από τα θετικά αποτελέσματα και όπως είπαμε και στην ε, Συμφωνία Πλαίσιο θα ξεκινήσουμε μια εντατική φάση δομημένου διαλόγου για τις μελλοντικέ πολιτικές προτεραιότητες μας. Η Κομισιόν αναμένει αυτές τις συζητήσεις και την ικανότητα να προωθηθεί μια καλύτερη σύγκληση Στην συνεδρίαση μας λοιπόν του Οκτωβρίου θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε έναν απολογισμό πριν την υιοθέτηση του προγράμματος. Τελικά όμως η επιτυχία αυτής της ατζέντας εξαρτάται από τη συνεργασία ανάμεσα σε Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Κομισιόν. Από τη γρήγορη προόδο στις πολιτικές διαβουλεύσεις και από την ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας επιτόπου στα κράτη-μέλη. Μόνο όταν δρούμε από κοινού και αποφασιστικά μπορεί η Ευρώπη να έχει τα αποτελέσματα τα οποία αναμένουν οι πολίτες, οι εταιρείε μας και οι επιχειρήσεις μας. Σήμερα λοιπόν κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστώ για την εξήγηση αυτή του προγράμματος και ζητώ συγγνώμη για το ότι ε, ο αποχαιρετισμός ε, του κυρίου Χριστόφια εξελίχθηκε σε μία μήνυ φωτογράφηση και ίσως ε, σας απέσπασε την προσοχή. Θα δώσω τώρα τον λόγο στον κύριο Ζωζεφ Σάιερ για τον για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που σας βλέπω στη θέση και του Πρόεδρου. Κύριε Αντιπρόεδρε Σεύκοβιτς, το μήνυμα του ΕΛΚ που συζητά το πρόγραμμα εργασιών του 2013 είναι σαφές και δείχνει ότι αυτό που θέλουμε να αφήσουμε για την επόμενη γενιά των Ευρωπαίων δεν είναι χρέη αλλά εργασίες, τις εργασίες και ευκαιρίες και δυνατότητες να προχωρήσουν. Όπως λέμε η Ευρώπη επί μακρόν ζούσε πάνω στο χρέος. Είναι ευκολότερος τρόπος να δαπανά κανείς τους πόρους και τα χρήματα των μελλοντικών γενεών και θα πρέπει να σταματήσει αυτό στην Ευρώπη για να δώσουμε κάποια ευμάρεια στις μελλοντικέ ε, γενιές θα πρέπει η Ευρώπη να βασιστεί στην εργασία εκ νέου και όχι στο χρέος και στις δυνατότητες θέσεων απασχόλησης. Σε αυτό το πλαίσιο η δυνατότητα να έχουν δουλειά οι νέες γενιάς και να μπουν στις αγορές εργασίας είναι ένα από τα σημαντικότερα μέτρα που συμπεριλαμβάνεται ε, στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά θα τονίσω εκ μέρους του ΕΛΚ ότι θα έπρεπε να είναι υπαριθμονένα ένα η προτεραιότητα αυτή. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την ανεργία των νέων. Φανταστείτε εκείνους που ξεκινάνε τη ζωή τους χωρίς να έχουν καμία προοπτική, καμία δυνατότητα να εργαστούν. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Θα πρέπει να δίνονται δυνατότητες στους νέους. Δουλειά να δώσουμε στους νέους και γι' αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Θα πρέπει και το περιμένουμε από το νομοθετικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτό να θέσουμε χρονοδιαγράμματα και στόχους σαφείς όσον αφορά την κινητικότητα των νέων, τις γλωσσικές γνώσεις και τα θέματα μαθητείας κλπ. Να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε ότι αυτό είναι περισσότερο έργο των κρατών μελών. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση με την νομοθεσία της θα πρέπει να βοηθήσει. Πολύ συχνά καυχόμεθα λέγοντα ότι έχουμε ελεύθερη κυκλοφορία όσον αφορά τα αγαθά υπηρεσίες κεφάλαια και άτομα αλλά λησμονούμε τα πάμπολα εμπόδια που εξακολουθούν να εμποδίζουν ε, τη δυνατότητα εφαρμογής αυτών των ελευθεριών, κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών. Το ΕΛΚ ζητά την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Θα πρέπει να αποκατασταθεί εμπιστοσύνη μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων σε αυτόν τον τομέα και εκεί υπάρχουν πολλές ε, νέες δυνατότητες. Επίσης, βασικό μας έργο είναι να μειωθεί η γραφειοκρατία, να δώσουμε καλά παραδείγματα στα κάτι μελη αλλά ε, να το πετύχουμε αυτό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να μειώσουμε το ε, γραφειοκρατικό άχθος από επιχειρήσεις και πολίτες. Αυτό το είδαμε και στο πρόγραμμα εργασιών αναφέρεται και στην πρότασή μας μείωση 25% μέχρι το 2015. Κάθε χρόνο Συνάδελφοι, συζητούμε το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και καμιά φορά αισθανόμαστε και το λέω επανειλημμένα κάθε χρόνο καμιά φορά αισθανόμαστε ότι είναι ένα μάταιο εγχείρημα διότι σύμφωνα με τις μελέτες μόνο κάτι λιγότερο το 50% των στόχων εμφανίζονται στις προτάσεις του επόμενου έτους από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ θα πρότεινα στην Επιτροπή ΑΦΚΟ να ετοιμάσει μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας που θα αναφέρεται στο πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό το ποσοστό. Δεν είμαι κατά της ευελίξιας. Κυρίως σε μια εποχή κρίσης θα πρέπει να υπάρχουν γρήγορες αντιδράσεις. Αλλά λειτουργεί ένα σχέδιο αν υλοποιηθεί. Αν δεν υλοποιηθεί ή υλοποιηθεί λιγότερο από το ίμιση, δεν πετυχαίνει τα βέλτιστα αποτελέσματα, άρα θα πρέπει να συνεργαστούμε για να τα βελτιώσουμε όλα αυτά. Εμπιστεύομαι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θεωρώ ότι είναι η δύναμη σταθεροποίηση τη θεσμικέ δομέ Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και αυτό αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολύ συχνά τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα κατηγορούνται ότι ακολουθούν τα γεγονότα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα, το δυναμικό, όλα τα μέσα για να ηγηθεί τη διαδικασία και σε εποχή κρίσεω ε, να μην ε, δείχνει τον δρόμο προ το μέλλον και μόνο, αλλά είναι και σημείο αναφορά και σημείο σταθερότητα εκ μέρου του ΕΛΚ, εκ μέρου του κόμματό μου και εκ μέρου του Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτού του είδου τη δραστηριότητα και να αυξήσουμε τη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Δεν ζηλεύουμε τη σχέση μεταξύ άλλων θεσμικών οργάνων, όπω με το Συμβούλιο είναι καλύτερε. Η Ρεμπέκα Χάρμ επέκρινε χθε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξέφρασε κάποια ζήλια γι' αυτό, αλλά εμεί δεν έχουμε πρόβλημα. Είμαστε ικανοποιημένοι αν σχέση μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι και αυτέ καλέ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σάιερ. Για του Σοσιαλδημοκράτε. έχει το λόγο ο κύριος Γκερέρο Σαλόμ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Στη χθεσινή συνεδρίαση ολομέλεια ζήσαμε μια σπάνια εμπειρία σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Υπήρξαν παρατεταμένες, παρατεταμένα συγγνώμη, χειροκροτήματα μετά την παρέμβαση του Πρόεδρου της Κομισιόν. Δεν είχε τυπικό χαρακτήρα, δεν είχε χαρακτήρα πρωτοκόλου ή οποιαδήποτε μορφή τέτοια. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει συνήθως να χειροκροτεί κανείς τον πρόεδρο της Κομισιόν, αλλά αυτό έγινε για δύο λόγους. Καταρχήν γιατί αφορούσε τη στάση του ότι ήταν έτοιμος να υπερασπιστεί τα γενικά συμφέροντα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και το έδειξε στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της προηγούμενης εβδομάδας και ιδίω έναντι των εκπεφρασμένων συμφερόντων πολλών κρατών, πολλών αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Αυτή η στάση λοιπόν ήταν κάτι το οποίο το εξετίμησε και ο πρόεδρος Σούλτς και όλο το κοινοβούλιο μας ή τουλάχιστον η συντριπτική πλειοψηφία των ε, βουλευτών και των Ευρωπαίων πολιτών. Επίσης όμως χειροκροτήθηκε ο κύριος Παρόσο γιατί υπήρξε μια κοινή αντιμετώπιση από, το, από την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο. Υπήρξε η κοινή ανησυχία των δύο αυτών θεσμικών οργάνων για την διάβρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της οικονομικής κρίσης που δημιουργεί προβλήματα στους πολίτες και ένδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει η ανησυχία αυτή γιατί αναδύεται και ενισχύεται ο ευρωσκεπτικισμός. Γιατί ενισχύονται οι ακραίες κατευθύνσεις και οι πολιτικές παρατάξεις οι σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει επιπλέον η ανησυχία για την υποβάθμιση των θεσμικών σχέσεων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο βλέπουμε να μας απογυμνώνει το Συμβούλιο από πολλές από τις αρμοδιότητές μας μέσω μιας πορείας προς τον διακυβερνητικό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τον αποκλεισμό της ενωσιακής μεθόδου από τη λήψη πολλών αποφάσεων τον τελευταίο καιρό. Πιστεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν ότι θα πρέπει να εργαστούμε από κοινού με την Κομισιόν για να προασπίσουμε τα συμφέροντα αυτά των Ευρωπαίων πολιτών. Θεωρούμε ότι πρέπει να εργαστούμε επίσης και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να υπάρξει μια κοινή λύση, μια κοινή λύση η οποία θα έχει υποστήριξη και προς την Κομισιόν και η οποία θα έχει μια κοινή πορεία με την Κομισιόν για να τηρηθούν τα στοιχεία αυτά που έχουν να κάνουν με την ενωσιακή μέθοδο. Το Κοινοβούλιο θέλει να υποστηρίξει την ανάπτυξη της θέσης απασχόλησης, την ευμάρεια, την ποιότητα ζωής, να επαναφέρει την εμπιστοσύνη των πολιτών μας. Θέλουμε μια καλύτερη οικονομική διακυβέρνηση, ένα καλύτερο δημοσιονομικό πλαίσιο προοπτικών, ένα καλύτερο ευρωπαϊκό ταμείο για την απόσβεση του χρέους, ένα οδικό χάρτη για τα ομόλογα σταθερότητας, καταπολέμηση της απάτης, ενίσχυση του ευρωπαϊκού ε, εξαμήνου και ένα καλύτερο επίπεδο πιστώσεων πληρωμών για το 2013. Σας λέω κύριε Πρόεδρε ότι οι περισσότερες πολιτικές ομάδες έχουμε αποφασίσει να αναβάλουμε την ψηφοφορία μέχρι το Σεπτέμβριο ώστε να υπάρχει περισσότερος χρόνος μέσα στον οποίο θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα κοινό ψήφισμα το οποίο να εκφράζει ομόφωνα, ενωμένα τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με τις απαιτήσει του και σε σχέση με την συνολική του υποστήριξη προς την Κομισιόν. Ευχαριστώ για τους φιλελευθέρους. Έχει το λόγο ο Άντριου Ντάφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι ένα πλούσιο πρόγραμμα για το 2013, το νομοθετικό πρόγραμμα της Κομισιόν και είναι πολύ σημαντικό γιατί αφορά το τελευταίο πλήρες έτος της ε, νομοθετικής εντολής του τρέχοντος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Κομισιόν έχει φτάσει πια στην κανονική της ταχύτητα λειτουργίας. Όπως αναφέρθηκε, χθες καταχειροκροτήθηκε ο κύριος Μπαρόσο και αυτό ήταν μια γνήσια εκδήλωση και μια πιστεύω σωστή και εύστοχη εκδήλωση από την πλευρά των ε, βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και έτσι αποστομώνονται και οι κριτικοί οι οποίοι οι οποίοι κατηγορούν συνέχεια την Κομισιόν ότι δεν είναι ένα εκλεγμένο σώμα, αλλά ένα σεσμός τεχνοκρατών. Εμείς ως φιλελεύθεροι πιστεύουμε ότι μια ισχυρή Κομισιόν πάντα πρέπει να θεωρείται ως μια πολιτική επιτροπή. Μπορεί να υπάρχουν φυσικά, να υπάρξουν κάποιες βελτιώσεις για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Κομισιόν υπάρχουν πολλές αρμοδιότητες και λειτουργίες της Κομισιόν και μερικές φορές ε, δεν είναι εμφανείς αυτές οι λειτουργίες. Καταρχήν η Κομισιόν είναι, είναι το πρόσωπο της Ευρώπης προς τον έξω κόσμο. Είναι επίσης ο διοικητικός μηχανισμός της Ευρώπης, ο οποίος θα πρέπει να είναι αποτελεσματικός και λειτουργικός και να έχει μια αποτελεσματική λειτουργία εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου. Επίσης, πρέπει να είναι η δεξαμενή σκέψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο χώρος προβληματισμού και οραματισμού για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να διερευνήσει και θα πρέπει να αρθρώσει καλύτερα και το κοινό συμφέρον των κρατών και των πολιτών που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν, αν χρησιμοποιήσει πλήρως και εκμεταλλευτεί πλήρως το δικαίωμα πολιτικής πρωτοβουλίας η Κομισιόν και ιδίως στις τωρινές συνθήκες που είναι ε, αντιμέτωποι με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτό θα είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κομισιόν αποδυναμώνεται όταν κρατάει αμυντική στάση, όταν γίνεται απλώς συνεργός αποφάσεων που λαμβάνονται και κλεισμένων των θυρών μεταξύ δύο ή τριών αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Η ισχύ της Κομισιόν προκύπτει από την δυνατότητά της να παραμείνει πιστή στο κοινό συμφέρον και να το προασπιστεί. Γι' αυτό χαιρετίζουμε το χωρίς προηγούμενο αυτό έγγραφο το οποίο διατυπώθηκε από τους τέσσερις προέδρους και το οποίο προτείνει ένα, ένα σχέδιο, μια ηλιοτυπία, ένα οδικό χάρτη για την μεταρρύθμιση στον τραπεζικό, στον δημοσιονομικό αλλά και στον πολιτικό χώρο στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Για τους πράσινους η κυρία Τούρουνεν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλω να πω ότι είναι σαφές ότι η κρίση θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο των πολιτικών που θα ακολουθήσουμε το 2013, διότι αν δεν καταφέρουμε να επιφέρουμε τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, θα παραλύσουμε στη χειρότερη περίπτωση ή θα διαλυθούμε ακόμα χειρότερα. Οπότε χρειάζονται οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις, σηματοπιστωτικές βραχυπρόθεσμα, αλλά και οι μακροπρόθεσμες θεσμικές αλλαγές θα πρέπει να έχουν πολύ υψηλή ε, προτεραιότητα. Και οι σχέσεις μεταξύ κρίσεως και του προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να είναι δυναμική σχέση. Διότι κρίση σημαίνει ότι ε, δεν είναι μόνο μία ετήσια απέτηση για προσαρμογέ, αλλά και εβδομαδία πρέπει να γίνονται προσαρμογέ. Δεν πρέπει να περιμένουμε το 2013 να ξεκινήσουμε με τα τέσσερα αυτά πακέτα μέτρων, το πακέτο τεσσάρων μέτρων. Θα πρέπει να εφαρμόζουμε πολιτικές αντιμετώπισης κρίσης. Αλλά όχι μόνο αυτό, κοινωνικές και ε, περιβαλλοντικές πτυχές ε, θα πρέπει να έχουν υψηλή προτεραιότητα όσον αφορά την ανάπτυξη. Χρειάζεται οριστική προσέγγιση για τη μετώπιση της κρίσης. Αυτή είναι η μόνη βιώσιμη λύση. Και θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα όσον αφορά το Ταμείο Αποπληρωμής του Χρέους στην Τραπεζική Ένωση ε, να υπάρχουν πιο συγκεκριμένες απαιτήσεις που καλύπτουν τις χώρες που παίρνουν κρατικές ενισχύσεις χρειάζεται μια εξυγίανση των τραπεζών χρειάζεται ε, αποκατάσταση των μακροοικονομικών ανισορροπιών ε, και οι χώρες οι πλεονασματικές και ελληματικές ε, να λύσουν τα προβλήματά τους ε, φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή, φορολογική παράδειση που να καταποληθούν να επιβληθεί φόρο σχηματοστητικές συναλλαγές χρειάζεται καλύτερη προσέγγιση όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης να ληφθούν υπόψη όλοι οι στόχοι του 2020 θα πρέπει να προσπαθήσουν τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν ένα μέλλον για την νεολαία της Ευρώπης. Οι απομένουσες προτεραιότητες αναφέρονται στη γραπτή μας δήλωση και στο ψήφισμα της ομάδας μας. Θα ήθελα να πω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να είναι πιο ενεργή όσον αφορά την επιδίωξη των στόχων του 2012 και 2020. Ο Μάρκομ Χάρμπορ. Uh, ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ πως είναι απολύτως απαραίτητο το πρόγραμμα αυτό να το δούμε ως ε, την, τον ηγετικό ρόλο της Κομισιόν στον τομέα των αναπτυξιακών πολιτικών. Αυτό είπαμε εμείς και χαίρομαι για αυτά τα οποία είπε ο Ιωζεφ Σάιερ γιατί συμφωνώ πάρα πολύ μαζί του και είμαι απογοητευμένο, γιατί νόμιζα πω θα είχαμε συμφωνήσει στο ψήφισμα για τι αναπτυξιακέ πολιτικέ. αλλά συμφωνώ με τον Ιωζεφ Σάιερ πω μέρο του προβλήματο είναι πω έτσι όπω παρουσιάζεται το πρόγραμμα δεν δίνει κάπου καθαρό βάρος και έμφαση στους στόχους της ανάπτυξης και τους στόχους της Κομισιόν μάλιστα ανταποκρίνεται πάρα πολύ σε αυτό το οποίο ζήτησε η Επιτροπή μου δηλαδή να δώσει προτεραιότητα στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Η νομοθεσία περί εσωτερικής αγοράς είναι το πρόγραμμα το αναπτυξιακό του επομένου έτου. Δεν το αναφέρατε στο λόγο σα, αλλά εκεί είναι οι στόχοι. Έχουμε τι ολοκληρωμένε πολιτικέ που ζητούσε η κυρία Τούριναν. Οπότε αυτό το οποίο θέλουμε από εσά, κύριε Επίτροπε, είναι να παίξει ηγετικό ρόλο στην αναπτυξιακή πολιτική. Αν δείτε τώρα τι δηλώσει του Συμβουλίου, γιατί ε, ε η εσωτερική αγορά δεν θα προέλθει μόνο από τις πολιτικές κομισιόν αλλά από την εφαρμογή στα κράτη-μέλη. Αυτό το οποίο λοιπόν πρέπει να δούμε στο πρόγραμμα του 2013 είναι ένα πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη-μέλη μπορούν να δεσμευτούν για τα αποτελέσματα, για τις δεσμεύσεις στην κοινή αγορά. Αυτό υπάρχει τώρα στη δήλωση του Συμβουλίου, πως η Κομισιόν δηλαδή θα παρακολουθεί την απόδοση και θα έχουμε μία έκθεση προόδου. Αυτό είναι λοιπόν αυτό το οποίο αναμένουμε. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να τονίσω και πάλι συμφωνώ εδώ με τον κύριο Σάιερ είναι πως η Κομισιόν αυτή τη στιγμή είναι υπόλογη για την μείωση του διοικητικού βάρους και τα κράτη-μέλη. Είναι στο πρόγραμμα εδώ πέρα. Λέτε πως θα κάνετε μια ανακοίνωση στο τέλος του έτους για περαιτέρω βήματα. Αυτό το οποίο θέλουμε να δούμε είναι αποτελέσματα εντός του 2013. Και επιπλέον πρέπει να δούμε το πώς περνάει η πολιτική, πώς θα γίνει περισσότερη προνομοθετική δουλειά στο Κοινοβούλιο, καλύτερη ανάλυση, αξιολόγηση αντικτύπου. Αυτά περιμένουμε στο πρόγραμμά σας για την ανάπτυξη. Συμπερασματικά λοιπόν κύριε Πρόεδρε, θέλουμε να δούμε το βασικό ζήτημα το οποίο είναι αποτελέσματα, δουλειές και ανάπτυξη. Και όπως είπε και ο Ζωζεφ Σαΐρ, η ανάπτυξη έρθει από τις μικρές επιχειρήσεις στον τομέα των υπηρεσιών. Έχουμε την οδηγία των υπηρεσιών, εμείς, εσείς και τα κράτη-μέλη από κοινού πρέπει να οδηγήσουμε σε ανάπτυξη και δουλειές. Ευχαριστώ η κυρία Μαρτίνα Άντερσον. Ευχαριστώ. Ο Λία Μέλλο είχε πει για μια άλλη συνθήκη πως πέρασε όχι επειδή το ήθελε ο κόσμος αλλά επειδή ο κόσμος φοβόταν και η δημιουργία φόβου φαίνεται πως είναι η απάντηση των θεσμικών οργάνων της Ένωσης στις διαμαρτυρίες για την αποτυχημένη πολιτική της λιτότητας. Οπότε το πρόγραμμα της Κομισιόν πρέπει να προσφέρει μια νέα προσέγγιση να μπουν πρώτα οι ανάγκες των ανθρώπων πριν από τα κέρδη, να αναγνωρίσουμε πως τα μέτρα λιτότητας είναι, ε, πλήττουν ιδιαίτερως γυναίκες και παιδιά. Το πρόγραμμα πρέπει να προωθήσει τις δημόσιες επενδύσεις, τις δουλειές, την ανάπτυξη, να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να δει ιδιαίτερα τι ανάγκε του κάθε κράτου μέλους. Αυτή πρέπει να είναι η βάση οποιασδήποτε αξιόπιστη στρατηγική επίλυση της κρίσης. Θα ήθελα λοιπόν να πω, επειδή ο χρόνο πιέζει, πως χρειαζόμαστε κοινή γεωρική πολιτική ευέλικτη με ε, επαρκή χρηματοδότηση. Πρέπει να απορρίψουμε την, μακροοικονομικού όρου για πρόσβαση στην πολιτική συνοχή και τα Ταμεία ανάπτυξη, να υπάρξει εγγύηση νεολαία για καλές δουλειέ και εκπαίδευση και ένα νέο οδικό χάρτη για ισότητα για τα άτομα ΛΟΑΤ και βεβαίω την εφαρμογή των στόχων της ε, Βαρκελόνης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ υπενθυμίζω συναδέλφου πω συνεχίζεται η συζήτηση. Έχω ακόμα τρει ομιλητέ. παρακαλώ όσοι μπαίνουν στην αίθουσα να σεβαστούν τους ε, υπολείπους οι οποίοι θα μιλήσουν. Σα ευχαριστώ, κύριο Φρανκ Φανχέκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίω. μπορεί να είναι ευσεβή πόθη, αλλά η Κομισιόν ε, εδώ πέρα παρουσίασε ένα πρόγραμμα ε, όπου λέει πως θα πρέπει πρώτος στόχος να είναι ανάπτυξη και δουλειές. Εδώ πέρα πρέπει να πει με κούλπα. Γιατί βλέπουμε πως η κρίση πλήττει τη δική μας ήπειρο χειρότερα από τις άλλες ε, υπήρους. Παρόλες τις διάφορες υποσχέσεις που μας λέγατε πως θα έχουμε την πιο αποδοτική οικονομία του κόσμου. Όλα αυτά έχουν πάει στον κάλαθο των αχρήστων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν τι κάνει υπό αυτές τις συνθήκες. Μας λέει πως ε, το 2013 πρέπει να αυξηθεί ξανά ο προϋπολογισμός Ένωσης. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ο καθένας μας εδώ πέρα έχει δεκάδες αν όχι εκατοντάδες παραδείγματα σπατάλης χρημάτων από τα ίδια τα θεσμικά όργανα. Πέρα του ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια εξορισμού δεν ξοδεύονται το ίδιο καλά με τα εθνικά. Μιλάμε δε για νέα παντελώς άχρηστα, παντελώς άχρηστες αποκεντρωμένες υπηρεσίες και συμβουλευτικά όργανα, επιδοτήσεις, τεράστια ποσά που πάνε στην ευρώφιλη προπαγάνδα και τεράστιες πατάλες στην αναπτυξιακή πολιτική. Θα πρέπει η Κομισιόν να καταθέσει ένα πρόγραμμα με ουσία να πετάξουμε το έρμα για να οδηγηθούμε επιτέλους σε οικονομική ανάπτυξη για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ καθίστε. Σταματήστε σας παρακαλώ τα πηγαδάκια. Τον λόγο έχει ο κύριος Άντριου Μπρόνς. Ευχαριστώ. Και παραθέτω, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε μικρή ύφεση και αυτό θα πρέπει να είναι η πιο εξωφρενική και παραπλανητική δήλωση και δεν αντιμετωπίζει, δεν αντιμετωπίζει την δηλαδή. Στην Ελλάδα και στην Ισπανία είναι περίπου 50% η ανεργία των νέων και ήδη έχουν εξάγει τι ε, θέσει εργασία και τώρα και του εκπαιδευμένου και του ειδικευμένου εργαζομένου. Η, Ευρωζώνη δεν αφήνει τι χώρε να αντιγωνιστούν κανονικά μέσω μειώνοντα το νόμισμά του. Μπορούν μόνο μέσω ε, λιτότητα να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και περιμένουν τι χώρε με τα μειωμένα εισοδήματα να βγουν από το χρέο. Η ελευθερία τη διακίνηση των εργαζομένων μεταξύ των διαφόρων χωρών που έχουν διαφορετικά επίπεδα αμοιβών άφησε ε, στη Δύση του ε, άνεργου του ε, εργαζομένου που δεν έχουν επαρκή δεξιότητα. Και στον Αμένο Βασίλειο αναγκάζονται να υπογράψουν σε διάφορα προγράμματα που δίνουν πολύ χαμηλέ αμοιβέ υπέρ των εταιριών. Και χώρε στην Ανατολή ταυτόχρονα έχουν στερηθεί του πιο ικανού εργαζομένου του με τα καλύτερα κίνητρα. Η μεγάλη απειλή η μεγαλύτερη απειλή για οδήποτε προσπάθεια για ανάπτυξη και απασχόληση είναι η παγκοσμιοποίηση και εμπορικέ συμφωνίε με αναδυόμενε οικονομίε με τι οποίε δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρεται στην επίτευξη μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Πραγματικό στόχο τη είναι ενιαία παγκόσμια αγορά, όπου οι αναδυόμενε οικονομίε και τα επίπεδα αυτών, αμοιβών αυτών, θα επιβληθούν σε όλου του εργαζομένου. Ευχαριστώ πολύ. κυρίε και κύριοι, είναι η ίδια κατάσταση όπως και χθε. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου σας ε, είπε, τον, είχε ήδη χθε ότι είναι πάντα προς το δικό μας συμφέρον να υπάρχει στο κοινοβούλιο μας ένα κλίμα το οποίο είναι το αρμόζον για την κοινοβουλευτική λειτουργία. Γι' αυτό σας παρακαλώ να καθίσετε και να ακούσετε την τελική παρέμβαση του Αντιπρόεδρου της Κομισιόν. Κύριε Σεύκοβιτς, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές οι οποίοι έλαβαν το λόγο εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή καταδεικνύει με σαφή τρόπο το ότι υπάρχει μια μεγάλη σύγκληση μεταξύ των σχεδίων της Κομισιόν για το νομοθετικό πρόγραμμα του 2013 και των προτεραιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως εκφράζονται μέσα από τις πολιτικές ομάδες. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε <clears throat> με αυτό το οποίο ανέφερε ο κ. Σάιερ ότι δεν πρέπει να αφήσουμε την επόμενη γενιά υπερχρεωμένη και χωρίς θέσεις εργασίας. Για Γι' αυτό τα μέτρα τα οποία προτείνει η Κομισιόν, τα μέτρα τα οποία θα εφαρμόσει η Κομισιόν είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να επιτύχουν αυτά τα αποτελέσματα τα οποία προσδοκούμε όλοι. Θέλουμε να τονίσουμε λοιπόν την ανάγκη να υπάρξει μια ευφυή εδραίωση στην οικονομία μα. Τα κράτη-μέλη μα θα πρέπει να απελευθερωθούν από το υπερβολικό άχθος χρέους, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει με έναν τρόπο ο οποίος δεν θα υπονομεύσει τις πολιτικές ανάπτυξη, που είναι οι πολιτικές οι οποίες δημιουργούν οικονομική μεγένθηση και θέσεις απασχόλησης. Αυτό πιστεύω ότι έγινε είναι ανάγλυφο στις συζητήσεις που είχαμε και με τα κράτη-μέλη σε σχέση με το θέμα της οικονομικής διακυβέρνησης και στις συστάσεις της Κομισιόν αναχώρα. Μια άλλη προτεραιότητα η οποία κατεδείχθη είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας και ιδίω της ανεργίας των νέων. Δυστυχώς. Έχουμε 7,5 εκατομμύρια νέους οι οποίοι βρίσκονται στο κενό αυτή τη στιγμή. Δεν είναι σε προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ούτε έχουν θέση εργασίες. Γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα με 8 κράτη-μέλη για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό και έχουμε ήδη συγκεκριμένα αποτελέσματα εκεί. Πάνω από 7 δισεκατομμύρια Κοντιλίων τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν χρησιμοποιηθεί για το στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόληση. Πιστεύουμε λοιπόν ότι με τα χρήματα αυτά θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε 460.000 νέε θέσει εργασία για του νέου άνεργου στην Ευρώπη. Για του άνεργου νέου μάλλον. Θέλουμε να μάθουμε από αυτή την εμπειρία και θα επεκτείνουμε το πρόγραμμα αυτό και σε άλλα κράτη-μέλη όπου παρουσιάζονται παρόμοια προβλήματα και πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος του ενεστώτος έτους θα μπορέσουμε να επανέλθουμε ενώπιον ημών με μια πρόταση για ένα κοινό πλαίσιο σε ό,τι αφορά την εγγύ... τις που θέλουμε να δίνουμε στους νέους ώστε οι νέοι να έχουν τη δυνατότητα να βρουν μια πρώτη θέση απασχόληση. Εγώ συμφωνώ με όλους τους ομιλητές οι οποίοι έχουν επιχειρηματολογήσει υπέρ της επιτάχυνσης των εργασιών μας για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Θα είναι αυτή η ψηφιακή αγορά ένα εργαλείο για δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ένα εργαλείο για την αύξηση του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η <clears throat> ταπεινή μας προσδοκία είναι ότι θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε μια αύξηση κατά 4% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2020. Πρέπει όλα αυτά να τα κάνουμε μαζί. Μας ενθαρρύνουν οι θετικές εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις μας για τους δημοσιονομικούς κανονισμούς έχουμε <clears throat> πράγματι υλοποιήσει την υποσχέσεις μας για τη μείωση του διοικητικού άχθους με στόχο να μειώσουμε κατά 30% μέχρι το τέλος του έτους και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν την ανάγκη αυτή απλοποίησης και την υπερβολική γραφειοκρατία. Συμφωνώ με τον Άντριο Νταφ και τον Ερήκε Σαλόμ όταν τόνισαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξασφαλίσει την προστασία των πολιτών. Ότι αυτό θα πρέπει να κάνουν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το σεβασμό της κοινοτικής μεθόδου και με τα σχέδιά μας για να υπάρξει μια σαφής τραπεζική, δημοσιονομική και εν καιρό πολιτική ένωση. Θα το πράξουμε λοιπόν αυτό όπως τόνισε η συνάδελφος από την ομάδα των Πρασίνων με μια ολιστική προσέγγιση και με μια βιώσιμη αντιμετώπιση. Για το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών έγινε σαφές στην τελευταία συνεδρία του ΕΚΟΦΗΝ ότι δεν θα έχουμε ομοφωνία για το θέμα αυτό. Η Κομισιόν λοιπόν θα προχωρήσει βαθμία εισάγοντας τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών μέσω της διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίας. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χάρμπορ για τις προτάσεις του για την πράξη της ενίας αγοράς και αυτά που λέει πρέπει να εφαρμοστούν και στη δεύτερη πράξη για την ενία αγορά είναι ένα από τα καλύτερα εργαλεία που έχουμε για να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για ανάπτυξη και δέσεις απασχόλησης. Και η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήθελαν να προχωρήσουν με ένα καλύτερο σχεδιασμό για την <clears throat> υλοποίηση των στόχων της ενιαίας αγοράς μέσα σε ένα πιο στενό χρονοδιάγραμμα μέσω της διαθεσμικής συνεργασίας. Αυτό θα μπορούσε να επιτύχει καλύτερη και ταχύτερη εφαρμογή αυτών των προτάσεων. Δυστυχώς δεν υπήρχε από την πλευρά του Συμβουλίου ο ίδιος ενθουσιασμός. Συνεχίζουμε όμως τις προσπάθειές μας για να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας στον τομέα της ενιαίας αγοράς. Για τα δύο τελευταία σημεία λοιπόν που αναφέρθηκαν, Έχουμε ήδη αναφερθεί στη σημασία του να έχουμε ένα σωστό πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για τη σημασία <clears throat> του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ένα σημαντικό εργαλείο και επίσης σε ό,τι αφορά τις εμπορικές πολιτικές μας. πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα σημαντικό εμπορικό εταίρος. Είμαστε μια μεγάλη εμπορική οντότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρέπει λοιπόν <clears throat> να λάβουμε υπόψη <clears throat> το ότι δεν έχουμε προχωρήσει σε επίπεδο μεγένθησης όσο οι εταίροι μα, οι Ηνωμένε Πολιτείες και η Ιαπωνία παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να αναπτύξουμε περισσότερο το εμπόριό μας με τους εμπορικούς εταίρους μέσα σε κοινά αποδεκτέ αρχέ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σας ευχαριστούμε πολύ για τις παρατηρήσεις σας αυτές για τη συζήτηση για το πρόγραμμα εργασίας κομισιών. Έχουν κατατεθεί έξι προτάσεις ψηφίσματος και πρέπει να ε, ψηφίσουμε για την αναβολή της ψηφοφορίας τον Σεπτέμβριο. Τελειώνει λοιπόν εδώ πέρα η συζήτηση και ξεκινάμε σε λίγη ώρα με την ψηφοφορία.